η παραμονή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίε. Καταρχήν θα ψηφίσουμε το αίτημα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αντίστοιχο αίτημα για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εξέταση σε δεύτερη ανάγνωση με βάση την απλωστευμένη διαδικασία της θέσης του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013. Δεν υπάρχουν ούτε τροπολογίες ούτε πρόταση απόρριψης, οπότε εγκρίνουμε την θέση του Συμβουλίου πάλι εξέταση σε δεύτερη ανάγνωση με βάση την απλουστευμένη διαδικασία της θέσης του Συμβουλίου για τους δείκτες κατανάλωση ενέργειας ε, και άλλων συνδεόμενων πόρων για ενέργεια ε, για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Δεν υπάρχουν τροπολογίε ούτε πρόταση απόρριψη, οπότε θεωρείται σε συγκεκριμένη πρόταση του Συμβουλίου, η θέση του Συμβουλίου. Και θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Μάνικα για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 1 του τρέχοντος έτους. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Εξετάζουμε τώρα την πρόταση ψηφίσματος και ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η έκθεση. με συγχωρείτε Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά που δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου. Θα έπρεπε να κάνετε κάτι, σας παρακαλώ. Καλώς, θα σας στείλουμε σωστικό συνέργειο. Παίρνουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Τσαρνέτσκι για την απαλλαγή 2008 του Γενικού Προϋπολογισμού. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαρνέτσκι. Κύριε Τσαρνέτσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε μια καλύτερη κατάσταση σήμερα από την πέρυσι, γιατί τότε την απαλλαγή την εγκρίναμε το Νοέμβριο. Φέτος έχουμε την ευκαιρία να την εγκρίνουμε αρκετά νωρίτερα, έξι μήνες νωρίτερα. Επιτέλους καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο να υποβάλει εγκαίρως ε, τα έγγραφα και μάλιστα πλήρως τεκμηριωμένα. Εμείς λάβαμε πολύ νωρίτερα τα έγγραφα φέτος και πιο ενημερωμένα. Και μάλιστα αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδήγησε στην ανάγκη άσκησης πίεση προς το, στο, Συμβούλιο για να αποκατασταθεί μια διαφάνεια για τα οικονομικά θέματα γιατί είναι απαραίτητη για να χορηγούμε την απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τσαρνέτσκι. Ε, ζήτησε το λόγο ο κύριος Μποντού. Το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί. Καλώς. Θα σας στείλουμε τεχνικό. Εξετάζουμε την πρόταση απόφασης για την απαλλαγή, χωρίς τροπολογίες. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκριση της απαλλαγής. Ε, την αναβολή θα, θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Όσοι θέλουν να δεχτούν την πρόταση για αναβολή της ε, ψηφοφορία απαλλαγή τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ. Όσοι δεν συμφωνούν θα ψηφίσουν κατά. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά για την πρόταση Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Τέλος. Απορρίπτεται η πρόταση. Ως εκ τούτου εγκρίνουμε την απαλλαγή. Περνούμε στην έκθεση Μικοβάσικ για τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Το λόγο είναι ο κύριος Μικοβάσικ. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Dnes je veľký deň. Deň Ευχαριστώ. Με την αποδοχή της οδηγίας αυτής καθιστούμε δυνατό να διασφαλίζεται η ποιότητα των μεταμοσχεύσεων. Παρακαλώ να υποστηρίξετε την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μικολάσικ. Έχουμε δύο μπλοκ τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε το πρώτο. Ποιο είναι υπέρ τη πρώτη δέσμη Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Περνάμε στη δεύτερη δέσμη τροπολογιών που καταπίπτει. Θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και θα ψηφίσουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος χωρίς τροπολογίες με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση. Θα ψηφίσουμε τώρα το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011. Το λόγο ο κύριος Φόξ, διαδικαστικό. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε κύριε Πρόεδρε ότι ψηφίζοντας την τροπολογία 4 θα μειώσει τον αριθμό επισκέψεών μας στο Στρασβούργο και ταυτόχρονα θα ε, μας επιτρέψει να τηρήσουμε την υποχρέωση της συνθήκης για 12 ολομέλειες το χρόνο στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, βλέπω από την λίστα ψηφοφοριών ότι προτίθεστε να θεωρήσετε μη παραδεκτή την τροπολογία 2. Παρακαλώ να ξανασκεφτείτε την αποφάση σας αυτή. Πράγματι, το 229 προβλέπει τις ε, περίοδου Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει όμως σχέση, δεν έχει μάλλον, ε, δεν βρίσκεται σε αντίφαση με την πρόταση της ε, πολιτική μου ομάδο. η οποία έχει το νόημα από την 10η εβδομάδα να μετατεθεί στην 11η εβδομάδα και δεν εμποδίζει να γίνεται την δεύτερη τρίτη του Μαρτίου μία ε, περίοδο συνόδου. Δεν υπάρχει μη παραδεκτό γι' αυτό. Σας παρακαλώ να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Λένε. Διαβάσετε τη σκέψη μου. Αυτό ακριβώς θα έκανα, αυτό που μαντέψατε. Ο κύριος Γκόλνης. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι παρά την αμφίσιμη σύνταξη, η τέταρτη τροπολογία θα έπρεπε να κηρυχθεί παρα, παραδεκτή, απορριπταία, διότι να γίνει μη παραδεκτή διότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου που προβλέπει την ε, διατήρηση του αριθμού των συνόδων στο Στρασβούργο στον ίδιο αριθμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι συνάδελφοι διαφωνούν. Η συνθήκη πάντως είναι απόλυτα σαφής και η απόφαση του δικαστηρίου με τη σημερινή νομολογία επίσης είναι απόλυτα σαφής. Καλώς. Ας ψηφίσουμε. Πριν ψηφίσουμε όμως, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η Προεδρία θεωρεί ότι η τροπολογία 2 δεν συνάδει με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος κρίνει μη παραδεκτή την τροπολογία 2. Το άρθρο 229 το άρθρο 229 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και σας διαβάζω το άρθρο, θα ε, συνεδριάσει χωρίς ανάγκη προηγούμενης σύγκλησης ε, τη δεύτερη τρίτη του Μαρτίου. Η συνδιάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε μία πρόταση χρονοδιογράμματος για το 2011 που προσθέτει μία ε, ολομέλεια 7 με 10 Μαρτίου τηρώντας με τον τρόπο αυτό το άρθρο 229 της, λειτουργίας, της Συνθήκης Λειτουργίας. Η τροπολογία 2 προβλέπει αναβολή αυτής της ολομέλειας για την επόμενη εβδομάδα, μετάθεσή της την επόμενη εβδομάδα. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την τροπολογία 2, θα παραβιάσει το άρθρο 229. Ως εκ τούτου θεωρείται μη παραδεκτή η τροπολογία 2. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμε. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα. Σωστά αναφερθήκατε στο άρθρο 229. Δεν βρίσκεται όμως σε αντίφαση με την τροπολογία μας. Το οποίο 229 αναφέρεται σε μία ημέρα του Μαρτίου, την δεύτερη τρίτη του Μαρτίου η τροπολογία μας αναφέρεται στην περίοδο συνόδου του Στρασβούργου στο σύνολό της, δηλαδή και στις τέσσερις ημέρες. Άρα πρέπει να είναι δυνατόν να μετατεθεί αυτή η περίοδος συνόδου από την δεκάτη στην ενδεκάτη εβδομάδα. Δεν απαγορεύει απολύτως τίποτα να γίνει μια ολομέλεια την δεύτερη τρίτη του Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Το προβλέπει όπως λέτε και η συνθήκη. Κύριε Ελένε, η τροπολογία 2 δημιουργεί πρόβλημα που θα, θα επιφέρει τελείως διαφορετικές ερμηνείες. Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ε, προβλέπει ότι τη τελευταία λέξη για την εφαρμοστέα ερμηνεία έχει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό και ο πρόεδρο κρίνει για του λόγου που σα εξήγησα ότι η τροπολογία 2 είναι μη παραδεκτή, γιατί κατά τη γνώμη μου παραβιάζει τη συνθήκη και συγκεκριμένα το άρθρο 229 τη συνθήκη. Φυσικά είναι σεβαστή οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Αλλά τον τελικό λόγο προβλέπει ο κανονισμό μα ότι τον έχει ο πρόεδρο. Και ο πρόεδρο κρίνει την τροπολογία 2 μη παραδεκτή. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Muy bien. Señorías, vamos a votar la... Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. κύριε και κύριοι, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καλώς. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ya está, si eh. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 3. Τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Se Τέλος. Απορρίπτεται η τροπολογία 4. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Τόσο κόντρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 1. Περάμε στο επόμενο σημείο. Ε, Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να επισημάνω στον Προεδρείο ότι θα πρέπει να παρέμβει, διότι οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Στρασβούργου και Ευρωπαϊκών Πρωτεύουσών θα πρέπει να είναι άμεσες, απευθείας και να μην δυσκολεύονται όσοι χρειάζεται να πάρουν τρει-τέσσερι πτήσει για να φτάσουν μέχρι το Στρασβούργο. Είναι μια έκκληση αυτή για να παρέμβετε και να ληφθούν τα μέτρα που χρειάζονται. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Σαλάτο. Seguimos. Pasamos a Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος με θέματα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. Το λόγο έχει ο κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μπορούμε να αποφασίσουμε ευθύ αμέσω. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος συστήνει στην Ολομέλεια να απαγορεύσει το κόλλημα τμήματων, κομματιών κρέατος ώστε να εμφανίζονται σαν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι, steak πρέπει να είναι steak. Το χειρομέρι να είναι χειρομέρι. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι ψηφοφόροι αυτό θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν υπερψηφίστε την πρότασή μας να απαγορευτεί η θρομβίνη ως πρόσθετο στα τρόφιμά μας. Muy Η ε, κυρία Γιούσο. Κυρία Γιούσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η θρομβίνη είναι ένα πρόσθετο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έχει κολλητική χρήση κολλάει τα κομμάτια κρέατος μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε τεχνολογικό ούτε ασφάλειας τροφίμων για τη χρήση της. Και μάλιστα τη χρησιμοποιεί τη θρομβίνη σε πολλές χώρες. Εγώ σας άκουσα, παρακαλώ ησυχία και εσείς για να με ακούσετε. Η πρόταση τροπολογία του παραρτήματο λέει ότι το κρέα που τη χάνει επεξεργασία με χρήση θρομβίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσυσκευασμένο με ετικέτα. Κάτι που δεν παραπλανάει, που δεν είναι το καταναλωτή. Γιατί αυτό θέλουμε να αποφύγουμε με το ψήφισμα, την παραπλάνηση του καταναλωτή. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο. Μήπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δεσμευθεί ότι προϊόντα που περιέχουν θρομβίνη να μην θεωρούνται ως απομιμήσεις κρέατος χάρη στην σωστή σήμανσή τους και μάλιστα ιδιαίτερα στα πλαίσια της αναθεώρησης του σχεδίου κανονισμού για την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τη διατροφή που προσφέρεται προς τον καταναλωτή. Θέλουμε να αποφύγουμε τις απομιμήσεις. Ο κύριος Επίτροπος. Well, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, βουλευτές. Η εξουσιοδότηση για το πρόσθετο της Τρομβίνης και μετά από συνεργασία της Επιτροπής με μέλη Σκεφτήκαμε τέσσερις προποθέσει, οι οποίες αναφέρονται και στον κανονισμό για τα πρόσθετα των τροφίμων. Αυτά είναι οι πτυχές της ασφάλειας, δηλαδή εάν υπάρχει σοβαρός τεχνολογικός λόγος, ή ανάγκε ενημέρωσης, τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη για τον καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε το τρόφιμο αυτό και αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του προσθέτου αυτού. Από την άποψη τη υγιεινή, λοιπόν, δεν μπορώ να συμμεριστώ την άποψη ότι σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνο μόλι είναι μεγαλύτερο από με άλλα προϊόντα. Όπω με το κρέα που, έχει περάσει, που έχει γίνει και εμάς οι τεχνολογικοί λόγοι που έχουν καταρτιστεί είναι ότι το προϊόν αυτό λειτουργεί ως σταθεροποιητικό για το τελικό προϊόν. Αυτή η τεχνολογική λειτουργία ρητός αναφέρεται στον κανονισμό για τα πρόσθετα των τροφίμων, ο οποίος υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Κατά τρίτον, οι πτυχές της ενημέρωσης Πρέπει να πω εδώ ότι μεγαλύτερε ανησυχίε που εκφράστηκαν στην έκθεση, ότι το προϊόν αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή, Μα οδηγεί στι εξή σκέψεις, ότι για να αποφύγουμε ένα τέτοιο κίνδυνο προτείνουμε ακριβώ τις εξή αυστηρέ προδιαγραφές, οι οποίες συμπτωματικά πηγαίνουν πιο μακριά από ό,τι συνήθως απαιτείται για τα πρόσθετα τροφίμων. Πρώτον, το προϊόν μπορεί μόνο να απολυθεί προσυσκευασμένο στον τελικό καταναλωτή. Δεύτερον, το προϊόν πρέπει να έχει επιπλέον ετικέτα που να λέγεται ότι πρόκειται για συνδυασμένα τμήματα κρέατος. Αυτό πρέπει να είναι πολύ κοντά στο όνομα τη εταιρεία πώληση. Ο καταναλωτή λοιπόν θα είναι πολύ καλά πληροφορημένο για την ακριβή φύση και την υφή του προϊόντο. Τρίτον, το όνομα του ενζήμου και τη προέλευσή του πρέπει να κατονομάζεται καθώ και η προέλευση και τα συστατικά. Να τονίσω ότι αυτέ οι απαιτήσει ετικετοθεσία είναι πιο αυστηρέ από ότι οι απαιτήσει που ισχύουν για άλλα προϊόντα με άλλα συστατικά όπως οι πρωτεΐνες αίματος και τα εγκεκριμένα προσθετικά, που έχουν ε, και αυτά επιπλέον απαιτήσει. Όμως εκεί δεν έχει απαιτηθεί η επιπλέον αυτή ετικέτα. Οι αυστηρότερες απαιτήσει ετικετοθεσίας θα είναι κάτι που θα το σκεφτούμε για το μέλλον. Τώρα η προετοιμασία αυτή του ενζήμου έχει ήδη μελετηθεί σε διάφορα κάτι μέλη ως ε, ένα μέσο για την ε, ε, καλύτερη προετοιμασία του προϊόντος. Εδώ τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να έχουν το χρόνο να, να κάνουν τις αλλαγές στην αντικαταθεσία που απαιτούνται ώστε να είναι καλύτερα ενημερωμένος ο καταναλωτής. Επίσης, οι καταναλωτές, ιδίως όσοι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, θα υποφεληθούν από την διάθεση φθηνότερων προϊόντων κρέατος, όπως και από την διαφορετική χρήση των διαφόρων τμήματων κρέατος κατά την επεξεργασία των ε, προϊόντων και του κρέατος γενικώ. Νομίζω ότι το συστατικό αυτό θα ωφελήσει και την αλυσίδα παραγωγής κρέατος και τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει λόγος για την εξάλληψή του και ελπίζω να καταλάβετε τους σοβαρούς αυτούς και ικανούς λόγους που σας περιέγραψα για να μπορέσετε να εγκρίνετε την πρόταση. Έχω δεσμευτεί προς το Κοινοβούλιο. Δεν θα πω σε κανέναν τι να καταναλώσει. Θα του εξηγήσω όμω τι είναι αυτό που καταναλώνουν, τι είναι αυτό που τρώνε. Και ακριβώ η θέση μου αυτή την κατοπτρίζει τη δέσμευσή μου. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματο. Απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία και ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση. Ψηφίζουμε την έκθεση Περεγιό για το σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Ψηφίζουμε καταρχήν το σημείο 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανείς δεν βλέπω να σηκώνει το χέρι. Παρακαλώ, ψηφίζουμε το τμήμα 4. Ποιος είναι υπέρ. Παράγραφος 4. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την παράγραφο 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία για την παράγραφο 4. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σε δύο τμήματα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 13. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της, της παραγράφου 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Σε Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23. 22, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Μάλλον έχει εγκριθεί η παράγραφος 22, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 22. Τέλος. Απορρίπτεται η παράγραφος 22. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της παραγράφου 33. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την αιτιολογική σκέψη L. Σε Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη εν Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος. Και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση Χάουρεγγι για τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 ποιος είναι υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ολόκληρη την πρόταση ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, πρόταση ψηφίσματος πέντε ομάδων για τη διάσκεψη αναθεώρησης του καταστατικού της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα. Το λόγο έχει ο κύριος Χόουιτ που προτείνει προφορική τροπολογία για, το, για την παράγραφο 3. Έχετε το λόγο κύριε Χόουιτ. Στην τρίτη τροπολογία, Πρόεδρε, θέλω απλώς να αντικαταστήσουμε το note σημειώνει με welcome καλωσορίζει. Κανεί δεν έχει αντίρρηση με την προφορική τροπολογία του κυρίου Χόουιτ. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία Τρία με την προφορική αλλαγή του κυρίου Χόουιτ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11, εδάφιο 1. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά Εποχές, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 11, εδάφιο 4, η ομάδα των πρασίνων θα καταθέσει προφορική τροπολογία. Την έχετε λάβει όμως και γραπτός. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Ψηφίζουμε. 11 εδάφιο 4 με την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 21 με προφορική πάλι τροπολογία του κυρίου Χόουιτ. Την έχετε λάβει και γραπτός πάντως. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία Χόουιτ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε την παράγραφο 21. Ποιος είναι υπέρ με την προφορική τροπολογία. Κατά Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 με προφορική τροπολογία της κυρίας Λόχμπιλερ. Την έχετε λάβει και γραπτός. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία Λόχμπιλερ. Όχι, οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 2 με την προσθήκη της προφορικής τροπολογίας Λόχμπιλερ. ¿Cuántos tienen que ser? 40. No hay 40, sí. Sí, hay, hay. Yo no cuento 40, ¿eh? A ver, no se muevan porque tenemos que... Ακίνητη, γιατί πρέπει να σας μετρήσουμε. Ακίνητη παρακαλώ. Bien. La Απορρίπτεται η προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Σκέτη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ολόκληρο το σχέδιο ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Επεξηγήσεις ψήφου πριν τη διακοπή. Για τον διορθωτικό προϋπολογισμό, το λόγο έχει η κυρία Ντότς.